E, Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο. Παρακαλώ. Καθίστε. Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία εκλογής του Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος δεύτερη φορά. Εκλογή Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, καθίστε.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 επί τη βάση των διατάξεων υπαριθμών 13, 15 και 18 του κανονισμού που προβλέπει τα σχετικά με την εκλογή των αντιπρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει κάποιος συνάδελφος αντιπρόεδρος, ο ενδέκατος, αντιπρόεδρος ε, εξελέγει βουλευτής στο Εθνικό του Κοινοβούλιο, έλαβε καθήκοντα προέδρου της Βουλής της χώρας του, για τον Παύλο Οπότε χειρεύει τώρα η θέση εκείνη και η οποία θα πρέπει να καταληφθεί από κάποιον άλλον αντιπρόεδρο και γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην σχετική εκλογή. Ε, η υποψήφη εξή. Λάσλο Τούρκης. Και ο υποψήφιος αυτός αποδέχεται την πρόταση υποψηφιότητας. Αυτή είναι η μόνη υποψηφιότητα. Οπότε για αυτό το λόγο σας προτείνω να ψηφίσουμε διαβοής. Όπως προβλέπει το 13, 3 διάταξη του κανονισμού μας. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ερωτώ, μήπως κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ένσταση ή επιφύλαξη κατά τις εκλογές. Κύριε Τούντα, έχετε το λόγο. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σήμερα για πρώτη φορά νιώθω ντροπή που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά κάποιο αρνήθηκε την συνθήκη ειρήνευση του Τριανών μετά τον ε, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προτάθηκε και εξελέγει για μια τόσο σημαντική θέση στην Ευρώπη. Πάρα πολύ. Ε, τώρα αισθάνονται προσβολή. Διακόπτει ο πρόεδρο στην μητρική του γλώσσα. Και, αλλά δεν μεταφράζεται και δεν ακούγεται. Θα πρέπει, συνεχίζει ο μιλητή, όλοι να βοηθήσουμε στο όραμα αυτό που λέγεται μια μεγάλη ενωμένη Ευρώπη. Σας ρώτησα εάν συμφωνείτε, το είπατε δεν συμφωνείτε, επομένως θα πρέπει τώρα να ψηφίσουμε όπως προβλέπετε. Θα γίνει κανονική ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, και διεξάγουμε τώρα την ψηφοφορία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε όλοι τις κάρτες σας. Μπορείτε να τις ε, εισαγάγετε στη σχετική σχισμή. Κύριε Σφόμποντα, θέλετε το λόγο. Μα ενημερώνουν ότι ο υποψήφιο θέλει να κάνει μια δήλωση πρώτα. Δεν ξέρω, αν μπορεί να έχουμε ε, σπαλμένη ενημέρωση. Αλλά αν θέλει να κάνει μια δήλωση υποψήφιο, νομίζω καλό θα ήταν να του δώσετε το λόγο. Ο πρόεδρο. θέλει να πει ε, λίγα λόγια ο υποψήφιο να απευθύνει το λόγο στο σώμα. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σύντομη δήλωση θα κάνω σήμερα. Την έχω προετοιμάσει, θα ήθελα να την αναγνώσω. Είναι για μένα μεγάλη τιμή ο διορισμός μου, η εκλογή μου μάλλον ως ε, Προέδρου του Ευρωπαϊκού, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγνώμη, την υποστήριξη και την πρόταση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχω λάβει ύψη ε, στο παράσημο της ε, Ρουμανίας το Δεκέμβριο του 2009 ε, στην επέτειο της 20ης επαιτίου της πτώσης της δικτατορίας στη Ρουμανία. Άνθρωποι από διαφορετική εθνική προέλευση και θρησκεία στη Τιμισοάρα που τους είχε ενώσει το ΣΕΝΟΣ και το θάρρος διέτρεξα τον κίνδυνο και με κίνδυνο της ζωής του στράφηκαν κατά του καθεστώτος του Τσαουσέσκου. Σήμερα συνεχίζω τις προσπάθειές μου στο πνεύμα εκείνης της εποχής για να εκπροσωπώ τα συμφέροντα της χώρας μου ε, στη υποστήριξη των μειονοτήτων, των θρησκευτικών ελευθεριών και των ελευθεριών γενικότερα. Είμαι προσιλωμένος ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές και χριστιανικές αξίες και στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ιδιαίτερα μιλώ για την κοινότητα ε, που εκπροσωπώ εγώ, την Ουγγρική μειονότητα της Ρουμανίας και είμαι μέλος του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην ε, κοινοβουλευτική του ομάδα. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίοδο που ακολουθεί τη θέση ισχύ της συνθήκης της Σαββόνας φέρνει νέα πνοή και ε, στην ιστορία της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε για τη δήλωση αυτή. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. θα ε, δείτε στις οθόνες σας να εμφανίζεται το όνομα ε, του υποψηφίου. Αν θέλετε να ψηφίσετε υπέρ του υποψηφίου, προφανώς θα ψηφίσετε το ΣΥΝ. Υπάρχει το πλήν, υπάρχει η αποχή, τα γνωρίζετε αυτά, είναι όλα απλά και γνωστά. Και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού, ο υποψήφιος εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία. Θα ανοίξει λοιπόν τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, Δέκα sekund. Δέκα δευτερόλεπτα θα χρειαστούν ε, για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα στις οθόνες σας. Głosowanie jest otwarte. Λοιπόν, η ψηφοφορία έχει ως εξής. Ψηφίσατε όλοι καταρχήν. What is the problem? Uh, not working. Δεν λειτουργούν τα μηχανήματα.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 E, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ, προσοχή λίγο. Όπως γνωρίζουμε, η ψηφοφορία αυτή χρειάζεται διακριτικότητα. Και ψηφίζουμε υπέρ, κατά ή αποχή. και έτσι καταγράφεται και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και αυτό κάνουμε σε ε, υποθέσεις προσωπικής ψηφοφορίας. Λοιπόν, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Κολέγο, Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Μπορεί να είμαι ο μόνος ε, ε, εδώ που δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Βλέπω μηδέν, βλέπω ένα, βλέπω σταυρό. Δεν ξέρω εγώ, είμαι ο στοιχείο του εδώ. Πώ ψηφίζει εδώ υπέρ κατά αποχή. Βλέπει ένα μηδέν, ένα ένα, ένα χ. Τι είναι αυτό. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε ξεκάθαρα. Ο πρόεδρο. αν θέλετε να ψηφίσετε υπέρ, θα πρέπει να ε, βάλουμε τον Κέρσορα εκεί ε, που έχει το θετικό πρόσημο, το συν. Αν θέλουμε να καταψηφίσουμε θα πρέπει να πάμε στο πλήν και αν ψηφίσουμε αποχή πηγαίνουμε στο μηδέν. Πρέπει να μετακινήσουμε λοιπόν στο μηχάνημα το Κέρσορα. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα τεχνικής φύσεως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ε, Πρόεδρε, κύριε Σούλτς, ε, με κάθε μετριοφροσύνη θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Εκεί δίπλα σας κάθονται μια σειρά συναδέλφων υψηλά αμοιβωμένων ε, που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν για να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Εγώ έχω μια οθόνη εδώ που γράφει το Ευχαριστώ πολύ. Μετά, έχω τρία κουμπιά στο μηχάνημά μου επίσης, που σε ονομαστικές ψηφοφορίε τα πατάω. Το πρώτο λέει ναι, το δεύτερο είναι αποχή, το μεσαίο και το τρίτο λέει όχι. Σωστά τα λέω. Μάλιστα. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Αυτό τώρα τι σημαίνει αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Τοκές θα, θα πατήσουν το ναι. Εκείνοι που δεν θέλουν να το ψηφίσουν θα ψηφίσουν το όχι. Και εποχή όπως είναι η πολιτική μου ομάδα θα πατήσει το αποχή. Καλά τα λέω. Ευχαριστώ πολύ. Tak, proszę Państwa. Ja dokładnie to przed chwilą powiedziałem, proszę Państwa. Πρόεδρος, ακριβώς αυτό έλεγα προηγουμένως. Ε, για όλους όσοι ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ πρέπει να ψηφίσουν το συν, όσοι θέλουν να καταψηφίσουν το πλην και όσοι θέλουν να δηλώσουν αποχή θα βάλουν το μηδέν. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, παίρνω και πάλι το λόγο, αν επιτρέπετε, μετά από την ερώτηση που έκανε ο Μάρτιν Σούλτ και τη δική σα αφέστατη απάντηση που είναι αντίθετη με αυτά που μου λένε οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου. Που μου λένε ότι μπορώ να ψηφίσω ναι ή αποχή, αλλά όχι, όχι. Ε, δεν είναι καθόλου σαφέ. Ε, ζητώ συγγνώμη που παίρνω το λόγο, αλλά να έχουμε κάποια συνοχή. Παρακαλώ, απαντήστε μου με σαφήνεια, κύριε Πρόεδρε. Ε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, λέει ο Πρόεδρος, ψηφίζουμε υπέρ ή κατά ή απέχουμε σε μια τέτοια ψηφοφορία. Και το κατά όπως και η αποχή συνυπολογίζονται. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Αν κάποιος ψηφίσει όχι ή αποχή είναι το ίδιο στην πράξη. Θέλετε να σας το επαναλάβω. Ψηφίζετε. Είτε το ναι, συν δηλαδή το κουμπάκι που λέει συν και αν απόσχετε ή καταψηφίσετε την υποψηφιότητα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μετράνε μαζί αυτές οι ψήφοι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ θέλω την προσοχή σας. Ακούστε. Να ψηφίσουμε να προκύψει το αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις τρεις, τρεις ερωτήσεις. Μόνο τρεις ερωτήσεις. Γιατί βλέπω πάρα πολλά χέρια που έχουν ύψωθει ε, στο ημικύκλιο. Οπότε σας παρακαλώ τώρα να θεωρηθεί ότι τελειώνει η ψηφοφορία για να μην κάνουμε καταμέτρηση. Απλώς για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε λήξασα την ψηφοφορία. Να μην κάνουμε καταμέτρηση τώρα. Τρεις ερωτήσεις. Δεν μετράει τώρα. Τρεις, τρεις. Εσείς εκεί πέρα, στο βάθος. Θεωρώ, θεωρώ ότι κατάφορα παραβιάζεται τον κανονισμό λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαράδεκτη αυτή η μεθόδευση που γίνεται να μην καταγραφεί καθαρά ποιοι είναι υπέρ κατά και πι λευκό. Διαπιστώνουμε εδώ από το χειρισμό των κουμπιών ότι το κατά δεν καταγράφεται. Πρέπει να δώσετε εντολή να καταγραφεί ξεκάθαρα η ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά και λευκό. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επομένη ερώτηση δεν είναι και τόσο δύσκολο να καταλάβει κάποιο ευφύς άνθρωπος ότι θέλουμε να ψηφίσουμε υπέρ, να ψηφίσουμε κατά και να ψηφίσουμε ω συνήθω και την αποχή. Δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε αυτό, γιατί αν δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε να μην ψηφίσουμε. Και η τρίτη ερώτηση τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας κάνω μια τεχνική παρατήρηση. Εδώ σε εμά το σύστημα λειτουργεί ως εξής. Πρώτα πατάς το ναι και μετά αν πας το όχι ακόμα μπλε είναι. Αν θέλεις να πατήσεις όχι δεν ανάβει τίποτα. Μόνο μέσω από το ναι περνά το όχι. Αυτά τεχνικά δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα. Ε, e, Κυρίες και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος, Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω, παρακαλώ την προσοχή σας, να έχει την καλοσύνη. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κυρία Ρότ. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο της. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, Ας τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα. Κανονικά, οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται στην αρχή της κοινοβουλευτικής ε, θητείας ε, και στο μέσον αυτής με βάση έναν κατάλογο. Εάν λοιπόν το κάνουμε αυτό και οποτεδήποτε γίνεται ε, μαθαίνει κανείς πόσες ψήφους, θετικές καταρχήν, πήρε στην άρφος και από εκεί προκύπτει και η σειρά που ε, διαμορφώνεται στο Προεδρείο. Σήμερα, επειδή προέκυψαν κάποια γεγονότα, ψηφίζουμε εκ των υστέρων για ένα συνάδελφο και αυτός χρειάζεται κάποιες ε, θετικές ψήφους για να εκλεγεί. Τίποτα άλλο δεν παίζει ρόλο, ε, συνάδελφοι. Η σημερινή εκλογή διαφοροποιείται από άλλες εκλογές. Η μυστική ψηφοφορία, αυτήν σας την περιέγραψε με απόλυτα η ακρίβεια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Πάτσα το σωστό κουμπί, βγήκε το μπλε φως και νομίζω ότι, εν περιπτώσει, όλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο που έκανα και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ πολύ ε, και συμφωνώ βεβαίως απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, εγώ προτείνω ε, σε ένα λεπτό ή τώρα, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε. Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ να ψηφίσουν το κουμπάκι για το υπέρ. Όσοι είναι κατά ή επιθυμούν να δηλώσουν αποχή, να πατήσουν το άλλο κουμπάκι. Όπως το εξήγησα την πρώτη φορά, δεν πρόκειται για κάτι το καινούργιο, το εξήγησα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. What is going on? Panie jest otwarte. Głosowanie jest otwarte. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ξανά. Proszę głosować. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Zamykam głosowanie. Τώρα ε, κλείνει, πέρασε τις ψηφοφορίες. 334 ψήφοι ζω. 3234 τέσσερις ή κατά 287 ογδόντα αποχές. Ο ε, αντιπρόεδρος μας. Ε, ε, έλαβε ειδική πλειοψηφία. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Λάσλο Τόκες που ε, συγκέντρωσε τις ψήφους που του αρκούν για να εκλεγεί αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του ο κύριος Αντιπρόεδρος Τόκες θα είναι ενδέκατο στην τάξη ε, μεταξύ των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Well, three, three, one. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου και η κάρτα μου και θα ήθελα να ληφθεί υπόψη. Ε, Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, πάρα πολύ που είμαι αναγκασμένος ε, να παρατείνουμε τη διαδικασία, αλλά αυτό που είπατε στην αρχή ήταν ή να ψηφίσει κανείς υπέρ ή να δηλώσει αποχή. Και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει υπέρ, κατά και αποχές. Ε, εγώ θεωρώ ότι αν κάποιοι ήξεραν ότι υπάρχει αυτή η επιλογή θα ψήφιζαν διαφορετικά. Άρα δηλαδή θέλω να πω το εξή ε, Εάν αυτό είναι ο σωστό τρόπο, δηλαδή να μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ, κατά και εποχή να επαναληφθεί η ψηφοφορία για μία τελευταία φορά. Πρόεδρος, σα ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, όσον αφορά επιφυλάξει σε σχέση με αυτή την ψηφοφορία, θα αντιμετωπιστούν με την πεπατημένη. Εμείς ε, θα προχωρήσουμε με βάση την ειδική πλειοψηφία που συγκέντρωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Τεκές, ο οποίος ε, εξελέγει και όλες οι αντιρρήσεις θα ληφθούν υπόψη και παρακαλώ πάρα πολύ αν έχετε αντιρρήσεις ή διαμαρτυρίες να έρθετε να με βρείτε σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί και εγώ θα μπορέσω να απαντήσω στις αντιρρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. morning. just uh, Ωραία, επομένω κάνουμε επανεκκίνηση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Θα πάρει ένα-δύο λεπτά, αλλά ο κύριο Βόμποντα έχει ζητήσει και έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να σας κοινοποιήσω ότι σύμφωνα με την ψηφοφορία έχουμε 789 μέλη στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι λίγο πλεονασματικό. Ελπίζω στις επόμενες ψηφοφορίες να μην αθροίζουμε 789 βουλευτές εδώ μέσα. Oh, Για αυτό που είπε ο κύριος Σφόμποντα, ο πρόεδρος. Αν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε στο τέλος της ψηφοφορίας θα σας ενημερώσω. Σε Ρόμπερτ Άτκινς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σφόβοτα έχει απολύτως δίκιο ο καλός φίλος μου Μάλκομ Χάρμορτ άθρησε το αποτέλεσμα και ακόμα και αν ψήφισαν και απόντες φτάνουμε στο 785 έστω και 789 ακόμα και ενισχύει αυτό τότε οπωσδήποτε είναι άκυρη ψηφοφορία και αυτό που πρέπει να κάνουμε Και τι πρέπει να κάνουμε κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ επιγόντως να το θέσετε υπόψη του Προεδρείου μόλις φύγετε από την Προεδρία να επαναληφθεί αύριο η ψηφοφορία είτε με κάλπη και χαρτί είτε με ένα σύστημα που να λειτουργεί σωστά πριν το τέλος των ψηφοφοριών θα προσπαθήσω να σας αναφέρω. Φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά και ανάμεσα σε αυτά που μετρήσατε εσείς, Ρόμπερτ και ο κύριος ε, Δεν θέλω να το παρατείνω αυτό. Το θέμα πρέπει να εξεταστεί, εξετάζεται αυτή τη στιγμή και θα σας αναφέρω το συντομότερο. Να πάμε στις ψηφοφορίες τώρα γιατί θα μας πάρει καμιά ώρα. Το πρώτο θέμα τώρα είναι λοιπόν η έκθεση κυρίας Ματέρα Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πριν ψηφίσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, Μπάρμπαρα Ματέρα οι εξελιγμένε οικονομίε είναι το θέμα τη απασχόληση. Είναι μια απειλή που έχει λάβει ανησυχητικέ διαστάσει σε περίπου το 10% στην Ευρωζώνη. Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού του 2011 προβλέπουν μία σειρά μέτρων ε, για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη και μεταξύ αυτών την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Διεθνοποίησης και Παγκοσμιοποίησης. Εγώ λοιπόν είμαι συγκήτρια αυτού και υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για ε, λειτουργία αυτού του Ταμείου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να συσταθεί αυτό το Ταμείο με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα να δίδονται απαντήσεις στους εργαζόμενους τομέων που πλήττονται από την κρίση και στις περιπτώσεις εταιριών που με μετεγκαθίστανται. Θέλουμε λοιπόν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ονομαστικά τώρα, αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. The vote is closed. Πέρας. εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ, 25 ε, αποχές και 51 κατά. Επόμενη ψηφοφορία και πάλι ονομαστική είναι έκθεση της κυρίας Ματέρα πάντα. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και πάλι. Επόμενο θέμα, πάλι της κυρίας Ματέρα, πάντα για την κινητοποίηση του Ταμείου. Ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται επίσης. Και επόμενη έκθεση, τέταρτη της κυρίας Ματέρα. Και πάλι ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται επίση. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Τρεμόπουλου διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηματοδότησή τη. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πριν την ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριε Τρεμόπουλε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κίνητρο για αυτή την έκθεση για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης επιτρέπει τη συμμετοχή πολιτών σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. η έκθεση αυτή που μου ανατέθηκε από την επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης περιέχει συστάσεις πώς θα πρέπει να περιληφθούν σε μελλοντικού κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία όπως η παροχή επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων και οι επαρκώς δεσμευτικοί κανόνες για την εταιρική σχέση. Άλλε προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχή, είναι για παράδειγμα ο ορισμό εκ μέρου τη κομισιόν μια πιο λεπτομερού και περιγραφικής παρουσίαση που προσδιορίζει τη δομή τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιέχονται. ακόμη η σύνδεση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια με τους νέους δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο μια σκληρότερη γραμμή από τους ελεγκτές για τις απαιτήσει επικοινωνίας και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένης και της κατονομασίας και διαπόμπευσης και της χρήσης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απάτης μια στενότερη εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων συναφών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και εφαρμογής της συνοχής καθώς και πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου περισσότερη καθοδήγηση από την επιτροπή σχετικά με το πώς να τεθεί η ρήτρα εταιρικής σχέσης στην πράξη από προγράμματα και βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση των μεγάλων έργων. θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για το τελικό αυτό κείμενο που μπορέσαμε να επιτύχουμε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ψηφίζουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για την έκθεση του Τρεμόπουλου. The Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλε. Η επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Κέλλη. Χρηματοδοτικέ συνεισφορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνέ Ταμείο για την Ιρλανδία. Ο συγητή έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι δεν, ε, δεν τους αρέσει τους συναδέλφους να μιλάνε τώρα οι συγγητές. Λίγα λεπτά την υπομονή σας. Δεν συζητήθηκε αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Κυρίω για το ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ταμείο για την Ελλάδα θα πρέπει να μιλήσουμε όμω. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα και εκτό τη θα θεωρήσουν ότι η ΙΠΑ χρηματοδότησαν σε μεγάλο βαθμό το ταμείο αυτό και βέβαια έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο και τους ευχαριστώ και τον Καναδά και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από το 2006 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε 57% των πόρων του ταμείου και δεν είναι ευκαταφρόνητο αυτό και δεν είναι και ευρέω γνωστό. Δεν έχει γίνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο, το έχουμε κρατήσει μυστικό, αλλά ήθελα να τονίσω ότι διαδραμάτισε ρόλο η Ένωση και ήμασταν ε, και βοήθησε για το διάλογο, τη συμφιλίωση και την ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία. Την ευχαριστώ και ε, η ρευτική διαδικασία ισχύει ακόμα ε, παρόλο που είναι εύθραυστη. Και ευχαριστώ όλους εκείνους που συνεισέφεραν για την ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι πάρα πολλοί και ιδιαίτερα τα άκρα ε, κόμματα όπως το δόκτωρο Πέσλι που ήταν εδώ μέλος επί σειρά ετών, το κόμμα του Τζέρι Άνταμς που πριν από 20 χρόνια δεν θα ερχόταν ποτέ ε, σε διάλογο. Λοιπόν, τα δύο ακραία κόμματα ήρθαν στη τράπεζα του διαλόγου και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό και εμείς να της αποτίσουμε την τιμή που της αναλογεί. Και αυτό είναι το τίμημα της ειρήνης στη Βόρεια Ελλανδία. Ελπίζω να έχει συνεχιστεί η ειρήνη και ε, συνεχίζει στα Ελλανδικά ο κύριος και ελπίζω ομόφωνα να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους ε, που έπαιξαν ένα θετικό ρόλο στην ευτική διαδικασία στη χώρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι ψηφορία θα κάνουμε και ευχαριστούμε κύριο Κέλλη. Ψηφίζουμε τώρα.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 Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας ε, υπήρξαν άλλοι 150 επιπρόσθετοι ε, βουλευτές, οι οποίοι εντωμεταξύ εξαφανίστηκαν. Ίσως λοιπόν θα πρέπει κάποιος να το ψάξει κανείς αυτό το θέμα. Πού πήγαν αυτοί οι παραπάνω που ήταν εδώ και ψήφισαν για τον Αντιπρόεδρο. Όχι, δεν εξαφανιστήκαν και θα σας εξηγήσουμε ξεκάθαρα τι συνέβη όσον αφορά τον κύριο Τόκες. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι πρόκειτο περί παρεμβάσεως του Αγίου Πνεύματος. Ούτε καν σώμα μηχανή Θεού. Λοιπόν, κύριε Μαρινέσκο, θα ψήφουν την ε, δική σας πρόταση και τώρα το, ε, πρώτον ε, σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτη δέσμη διατάξεων. Πέρασε. Ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη δεύτερη δέσμη διατάξεων. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82 με χρωστή ψηφοφορία. Σε τρία τμήματα και τα τρία μονοκλή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Και τώρα, πρόταση του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, ναι, ευχαριστούμε και τον κύριο Μαρινέσκο και προχωρούμε τώρα στο κείμενο Μάρτιν. Ξεκινούμε με αυτή τη δέσμη τροπολογιών. Πώς είπατε, συγγνώμη, τι είπατε. Μάλιστα, σε Ρόμπερτ. Συγγνώμη που σα ενοχλώ και πάλι. Αλλά προβλέπετε εδώ και τέταρτη νομιστική ψηφοφορία σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουμε λάβει. Πρόεδρος. Από ό,τι μου λένε υπάρχει μια νεότερη εκδοχή των εγγραφών της ψηφοφορία. Επομένως αυτό που είπατε δεν ισχύει. Και θεωρείται λήξα σε ψηφοφορία επί της εκθέσεως Μαρινέσκου. Τώρα έχουμε 15 ψηφοφορίε από την Συνταγματική Επιτροπή επί τη εκθέσεω Μάρτιν και τι ψηφίζουμε τώρα ποιοι είναι υπέρ. Ναι, κύριε Γκέλνη. Διαδικαστικό. Γκέλνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνω ότι σε αντίθεση με τον κύριο Μπούζεκ δεν πάσχεται από πλάγιο στραβισμό και με είδατε. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχω ένα διαδικαστικό. Σύντομα, η έκθεση του κυρίου Μάρτιν φιλοδοξεί να ε, διορθώσει τα προβλήματα προσαρμογής συνθήκη της Σαββόνα. Αλλά μεταξύ των κειμένων που έχουμε να ψηφίσουμε υπάρχει ένα που δεν έχει καμία σχέση με τη συνθήκη της Σαββόνα και μου φαίνεται αντίθετο και με τις γενικές αρχές του κοινοβουλευτικού δικαίου. Είναι εκείνο που αφαιρεί από τους μη εγγεγραμμένου βουλευτέ τη δυνατότητα να ορίζουν μόνοι τους εκπρόσωπό τους. Ε, συνάδελφοι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές σας πεπιθήσεις, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ο πρόεδρος, όσο μερόληπτος κι αν είναι, να ελέγχει, να αποφασίζει με ποια κριτήρια θέμω άραγε Ποιο θα εκπροσωπήσει του μη εγγεγραμμένου στη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο αντιτίθεται στι Γενικέ Αρχέ Δικαίου και στην ομολογία του ΔΕΚ. Για το λόγο αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι η τροπολογία αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο ψηφοφορία σήμερα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mr. You may recall that for several months I sat as a non-attached member. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλνης. Μπορεί να θυμάστε ότι διατέλεσα επί σειρά μηνών μη εγγεγραμμένο μέλος και απέχουν τόσο πολύ απόψεις μου από τις δικές σας που αποδεικνύουν ότι μια εγγεγραμμένη ούτε είναι ούτε πρόκειται ποτέ να είναι κοινοβουλευτική ομάδα. 15 τροπολογίες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων τις ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μη 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 είπε. κατά αποχές εδώ χρειάζεται ειδική πλειοψηφία και έλεγχο συνεπώς. 121 αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία, επαλήθευση. check Πέρασε της ηλεκτρονικής επαλήθευσης. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε τροπολόγια παριθμών 2. Α, όχι, καταπίπτει. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Η δύο υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, να με συμπαθάτε. Λοιπόν, έχει καταπέσει, είπαμε. Τώρα, Περνάμε στην τροπολογία 96. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Όχι, καταπίπτει, συγγνώμη. Η 97 είπε Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 είπε Κατά. Αποχές. Έλεγχο σας παρακαλώ πολύ. 98 αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται 492 κατά 130 επέ. 99 επέ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο, αρχίζει για την 108. Ηλεκτρονική πολίτευση. Okay, τη check Εγκρίνεται. 396-250. Η 83 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. We now move to 112. Those in Υπέρ της 112 κατά αποχές εγκρίνεται. We now go to 62 to 64 together. 62 μέχρι 64 μαζί. Όχι, έχει καταπέσει λέει ο πρόεδρος. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180, 105 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, Λοιπόν, κύριε Μάρτιν, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ο εισηγητής. Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσω ε, την Ολομέλεια. Πριν ολοκληρώσουμε, έχω δύο τεχνικά ζητήματα, γιατί γνωρίζετε ότι η διαδικασία αυτή άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο. Θα πρέπει να προσθέσουμε μια νέα αιτιολογική αναφορά, για να συνδέσουμε ε, του Νοεμβρίου την ψηφοφορία με τη σημερινή και να λέμε, λαμβάνοντα υπόψη τη απόφαση του Νοεμβρίου 2009 για την προσαρμογή του κανονισμού του Κοινοβουλίου στη συνθήκη κτλ. Να προσθεθεί αυτή η αναφορά, είναι τεχνική και μόνο. Και το δεύτερο που είχα να πω, δεν μπορούμε να πουμε πρωτη Πρώτου 2009 να τεθεί σε ισχύ. Πλέον αυτό είναι ανέφικτο και θα ζητήσω να βρει εφαρμογή το άρθρο 201 εδάφιο 3, δηλαδή ε, την πρώτη μέρα μετά το πέρας της περίοδου της Συνόδου. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν για την ε, έκθεση αυτή και το έργο συνολικότερα. Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη έκθεση και δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα της συγγήτριας εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προεπλογισμού 2011. Ψηφίζουμε τροπολόγια 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Do you really want me to check Mr. Lambridge? I think he's joking. Um, I put amendments 1 and 18 to the vote by roll call. 1 και 18 ονομαστικά. Αρχίζει τώρα. The roll call is closed. Πέρας. Απορρίπτονται. Η 19 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ή 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 14 κατά τμήματα σε τρία τμήματα τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο, Υπε. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 και 21, ψήφι Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήταν σαφέστατο, δεν θέλετε έλεγχο. Υπε. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 17, κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο Είπε. κατά αποχές απορρίπτεται 15 Είπε. κατά αποχές απορρίπτεται η παράγραφο 46 Είπε. κατά δεν είναι πολύ σαφές αυτό θέλει έλεγχο αρχίζει για τη 46 Check is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στο 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ έλεγχος ηλεκτρονικός για την τροπολογία 25 πέρας εγκρίνεται απορρίπτεται απορρίπτεται 387 κατά 253 υπέρ ναι, ναι, από την πολύ βιασύνη έκανε λάθο. Σπέβδε βράδυ. 26 είναι υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5 και 28. Χωριστή ψηφοφορία. Και ονομαστική. Ψηφίζουμε. Για το πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Τροπολογίες 6 και 29 με χωριστή ψηφοφορία στις δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. και εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά έλεγχος για το 67. Check is closed. 490 in favor, 157 against. That was adopted. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά.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 Αποχές απορρίπτεται. Οκτώ. Έλεγχος για το οκτώ. Μου φαίνεται ότι ο πρόεδρος. Και ψηφίζουμε. Πέρας. I was wrong by margin of votes. It was a... Α, όχι, έκανα λάθος. Γιατί εγκρίνεται 326-319 και να με συμπαθάτε. Τροπολογία υπέρ 30. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με νομαστική ψηφοφορία. The vote is closed. And that's adopted by 571 45. Εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσμα με 571 ψήφου υπέρ, 45 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Το επόμενο. Έκθεση Λάγκεν. Όσον αφορά τα παράγωγα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 αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο K υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη S όπως sugar υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε για το ε, ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια κύριε Λάγκεν Τώρα ψηφίζουμε ε, για την έκθεση Μπαντία Κουτσέτ σχετικά με το διαδίκτυο και ίσως εδώ για αυτό το θέμα θα πρέπει να μας μιλήσει η για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Ε, θα ψηφίσουμε από κοινού για το 1 μέχρι 3 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνονται και τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της με ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια. Πάμε τώρα στην έκθεση Σόζα Βάγνερ για το ε, ίντερνετ των κυβερνήσεων, διακυβέρνηση του ίντερνετ μάλλον. Ψηφίζουμε για την έξι σε δύο τμήματα με ξεχωριστή ψηφοφορία και ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 6. Έκλεισε η ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 14. Επίσης με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγω 16 σε δύο τμήματα και τα δύο μονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται και αυτό. Πάμε τώρα στην παράγραφο 20. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 43. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία ε, Σόζα Βάγνε. Πάμε τώρα στην έκθεση Βίνκλα σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Ε, Παράγραφο 46 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 46, μάλλον με συγχωρείτε λέει ο λάθος, ε, για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βίνκλερ. Πάμε τώρα στην έκθεση Κάσμαν σχετικά με τους στόχους χιλιετίες. Πρώτη τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η επαλήθευση. Απορρίφθηκε με έξι ψήφους. 316 με 322 είναι το αποτέλεσμα. Παράγραφος 7. Ε, με ε, ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και αυτό εγκρίνεται. Πάμε τώρα για την παράγραφο 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Αν θέλετε, εντάξει, ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική επαλήθευση. Μέχρι τώρα τα πάμε πολύ καλά, λέει ο Πρόεδρος, από πλευράς χρόνου. Παράγραφος 8 παρακαλώ. Παράγραφος 8 άρχεται η επαλήθευση. Έκλεισε η επαλήθευση. Απορρίφθηκε 266 με 368. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Ε, ονομαστική ψηφορία, συγγνώμη, ναι. Ε, λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία ξεκινάει. Έκλεισε και απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά εν πάση άρχεται η, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε. Εγκρίθηκε 369 με 263 το αποτέλεσμα. Πάμε στην 22 ε, σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, ξεκινάμε, ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε. εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Άρχεται η... Ε, όχι, όχι, ε, δεν είναι ονομαστική ψηφορία. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 23. Σε δύο τμήματα ε, ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το δεύτερο. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε. Και απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η επαλήθευση. Εγκρίθηκε και ζητώ συγγνώμη. Είχα κάνει λάθος. 27. Υπέρ. Κατά αποχές ε, πολύ τσιματσίμα ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 27 την παράγραφο παρακαλώ έκλεισε η επαλήθευση η 27 εγκρίνεται παρακαλώ ε, κύριε Μπάσκεπα διαδικαστικό έχετε το λόγο Ζητώ συγγνώμη, εγώ ήθελα μόνο να πω ότι δεν λειτουργήσε η συσκευή μου. Μήπως μπορείτε να στείλετε τεχνικό, γιατί εγώ στην τελευταία ψηφορία δεν μπόρεσα να συμμετάσχω. Θα το πράξουμε αυτό, λέει ο Πρόεδρος, και πάμε τώρα στην παράγραφο 42 σε 4. Τμήματα για κάθε ένα από αυτά με ονομαστική ψηφοφορία. Για το πρώτο άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται Πάμε στο δεύτερο, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στο τρίτο τμήμα, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε για το τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την τροπολογία υπερθμών 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 47 με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη ε ή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη 6 υπέρ κατά επαν, επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται Πάμε τώρα ε, να ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος ε, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Και τώρα πάμε στην τελευταία ψηφοφορία και θα σας ε, ε, μιλήσω για την ε, περίπτωση για την εκλογή του Αντιπρόεδρου μετά την τελευταία ψηφοφορία. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάλι. Έκλεισε η ψηφοφορία, η ονομαστική ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Συγγνώμη, κύριε Κάσμαν, εγκρίθηκε το ψήφισμά σα. Συγχαρητήρια. Ε, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε εδώ στο Προεδρείο. Τώρα, το επόμενο θέμα αφορά στην ε, Επιτροπή την Κάρι Φόρουμ υπερκατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τώρα, συνάδελφοι, όσοι θέλουν να ακούσουν την εξήγηση για την ε, ψηφοφορία Τόκες, τα μέλη που ψήφισαν 621 και υπέρ και αποχές πάνε μαζί. Υπέρ 334. Αποχές 287. Η απόλυτη πλειοψηφία είναι 168. Ο κύριος Τόκες πήρε 333 ψήφους που είναι πάνω από την απόλυτη πλειοψηφία του 168. Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφορίας είναι εναλλακτική λύση ψηφοφορίας με την κάλπη. Όταν έχουμε την κάλπη μπορεί κανείς να ψηφίσει μόνο υπέρ και για συγκεκριμένο αριθμό ε, ψηφών. Δεν μπορεί κανείς να ψηφίσει κατά, όπως τα είπε και η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Όσοι δεν θέλουν να ψηφίσουν υπέρ, ε, ψηφίζουν λευκό. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαιρετίζω την εκλογή του κυρίου Τόκες στο Προεδρείο. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Κύριος Λαμπρινίδης, διαδικαστικό παρακαλώ. Mr. President, just... Κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβω λίγο.